Καλημέρα σε όλους. Ας αρχίσουμε. Έχω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις και μετά θα δώσω την προεδρία στην κυρία Βάιλερ, η οποία δέχτηκε να με βοηθήσει σήμερα το πρωί, γιατί εγώ έχω μια σύντομη συνάντηση εδώ έξω με τον νέο σύμβουλο του Βρετανού Πρωθυπουργού. Λοιπόν, Καλώς ήρθατε στις συνεδριάσεις μας σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα. Σήμερα το πρωί έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες και σήμερα το απόγευμα θα ανοίξουμε τη διαδικασία για διάφορα νέα θέματα. Το πακέτο για τα ταξίδια, ο κύριος Μάγερ είναι ο μας από το ΕΛΚ, και για την ενιαία αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που είμαι εγώ εισηγητής της Επιτροπής μας. Οπότε θα γίνουν παρουσιάσεις για αυτά τα δύο θέματα σήμερα το απόγευμα. Όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, έχω να σας πω ότι το σημείο 13 του κυρίου Χατζημαρκάκη αποσύρεται για την προσβασιμότητα σε ιστοσελίδες ε, του δημοσίου τομέα. Το μικρόφωνο μου πρέπει να το αλλάξω γιατί νομίζω ότι στο... για να φαίνομαι καλά στο web stream πρέπει να χρησιμοποιώ το αριστερό μικρόφωνο. Υπάρχει και ένα νέο news brief letter. Το δελτίο αυτό υπάρχει, είναι στη διάθεσή σας. Αν δεν το πήρετε στις θηρίδες σας, ευχαρίστω να σας το δώσουμε. Εξάλλου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το λαμβάνετε τακτικά. Θέλω επίσης, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Βάιλερ, να σας ενημερίσω όσον αφορά τι τριμερείς διαπραγματεύσεις, τον τριμερή διάλογο δηλαδή. Την Τρίτη καταλήξαμε σε συμφωνία με την Λιθουανική Προεδρία όσον αφορά το πρόγραμμα καταναλωτών 2014-2020. εκκρεμεί το ψήφισμα σχετικά με τον κοινοτικό προπολογισμό εδώ και αρκετό καιρό, η απόφαση γι' αυτό, οπότε γι' αυτό και εκκρεμούν διάφορα θέματα. Εμείς πάντως πετύχαμε τον έλεγχο όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων και την, στα μέσα του δρόμου αξιολόγηση, τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση για την κατάσταση πραγμάτων και εφόσον χρειαστεί να υπάρξει και μια νομοθετική προσαρμογή για να μπορέσει έτσι να προχωρήσει καλά το πρόγραμμα. Οπότε επιτεύχθηκε συμφωνία, θα επανέλθουμε βέβαια εδώ στην Επιτροπή μας ένα θέτο χρόνο για να ψηφίσουμε και μετά θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Είναι η διατροφική κρίση και οι αφάτες στην διατροφική αλυσίδα και ο σχετικός έλεγχος. Εμείς έχουμε γνωμοδότηση της κυρίας Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ, που είναι η συντάκτρια της νομοδότησης και επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος με την κυρία Ντελάνκερ, η συγγήτρια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους σκιώδους συγγητές που είναι εδώ. Συνεπώς, δίνω την προεδρία στην κυρία Βάιλερ και όταν φτάσουμε στις ψηφοφορίες θα έχω επιστρέψει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν βοηθάει να συζητήσετε με την Βρετανική κυβέρνηση. Είμαστε όλοι υπέρ να το κάνετε. Να μείνετε εκεί μέχρι να αρχίσουν οι ψηφοφορίε λοιπόν. Εντάξει. Συνάδελφε Κοράτσα Μπίλτ, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Uh, thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αλυσίδα, την τροφοδοτική, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους καταναλωτές. Νομίζω όλοι με την ίδια ανάλυση είδαμε τι συνέβη με το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο και με το αλογίσιο κρέας που δημιούργησε σύγχυση στους καταναλωτές. Και έχουμε ευθύνη από κοινού να βρούμε οδούς και τρόπους να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Προσπάθησα πραγματικά να λάβω υπόψη τις απόψεις σας και θέλω να ευχαριστήσω όλους που συνεισέφεραν με πολύ πολύ καλές τροπολογίες. Πρότεινα κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες από πλευράς μου και ελπίζω, ευελπιστώ ότι όλοι μπορούν ε, να συμπέσουν και να συμφωνήσουν σε αυτό το σημαντικό θέμα γιατί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Το αλογίσιο κρέας δεν ήταν θέμα ασφάλειας, τροφικής ασφάλειας. Ήταν ένα πρόβλημα παραπλάνησης στην ετικετοποίηση και στις συσκευασίες. Έδειξε η Επιτροπή ότι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και το σύστημα συντονισμού λειτουργήσε και η μη σωστή ετικετοποίηση οδήγησε στο να αφαιρεθεί αυτό από την αγορά, αυτό το στοιχείο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να βρούμε έναν τρόπο να προστατέψουμε τους καταναλωτές χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις και πρόστιμα για τις εταιρείες στο σύνορο της αλυσίδας που δεν είναι υπεύθυνε αυτές οι εταιρείες όλες για όλα όσα συνέβησαν. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει κάτι. Αν με πρόσθετη νομοθετική προσπάθεια, με πρόσθετες κυρώσεις και πρόστιμα χτυπήσουμε, πλήξουμε όλη την αλυσίδα, την τροφική, στο τέλος τέλος οι καταναλωτές θα πληρώσουν το κόστος και θα εξωθηθούν εκτός αγορών κάποιες εταιρείε που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Θέλω να πω ότι κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση, κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα, περισσότερο νομοθετικό έργο φαίνεται να είναι η μαγική λύση. Σε αυτήν όμως την περίπτωση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτική προσεκτικοί προτού προτείνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο και νέες νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε η υφιστάμενη κείμενη νομοθεσία να μπορεί να εφαρμοστεί και πλήρως να συμμορφώνονται όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτήν. Οι εγκληματίε που θέλουν να, απατήσουν πάντα θα βρουν τον πιο αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα και θα το κάνουν. Γι' αυτό τα τρία μέτρα που προτείνουμε είναι ένα καλύτερο ορισμό για την απάτη και γενικά για την ε, ε, τα θέματα τροφικής ασφάλειας. Πρέπει να αποσαφινιστούν κάποια πράγματα, διότι έχουμε κάποιες συγκεχημένες πληροφορίες μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας. Πρέπει όμως να μπορούμε να λειτουργούμε ακόμα και όταν υπάρχει απάτη ή ε, παραπλάνηση σε σχέση με τις ετικέτες, ε, τη συσκευασία και την ετικετοποίηση. Πρέπει να έχουμε και μελέτη ε, επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μελέτη βιωσιμότητας. Πρέπει να έχουμε την ε, των ετικετών για τα κρέατα ε, και να δούμε ότι το 50% για παράδειγμα για μια συστατική ουσία ε, γιατί διαφορετικά μια και ε, πολλές φορές υπάρχει θέμα με τους καταναλωτές και τις εταιρείες σημαντικό είναι να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμοσιμότητας και να μπορεί να ειχνηλατείται οποιοδήποτε στοιχείο ε, το οποίο εμπεριέχεται σε τέτοια τρόφιμα όταν είναι κρέας. Δεν νομίζω ότι αν είμαστε υπερβολικοί θα έχουμε ε, κάποια πρόσθετη αξία για τους καταναλωτές και δεν θα είναι όλα αυτά βιώσιμα και δεν θα είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Το τρίτο σημείο είναι η αύξηση των ελέγχων στο εθνικό επίπεδο. Φυσικά, καλύτερο συντονισμός, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών για την αντιμετώπιση των θεμάτων των τροφίμων, καλύτερες επιθεωρήσεις και έλεγχοι. Η έλεγχη όμως είναι και μια δαπάνη στοιχείο για τις επιχειρήσεις. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πρέπει να είναι αποτελεσματικές και αποτελεσματικές και όσον αφορά τις δαπάνες και να μην υπάρχει περιττό γραφειοκρατικό κόστος μόνο. Για τις ε, τροπολογίες το τρίτο ήταν τα πρόστιμα, οι κυρώσεις, το είχα ξεχάσει. <clears throat> Αυτή τη στιγμή ε, ίσως δεν λειτουργούν τα πράγματα αποτελεσματικά. Οι αστυνομικές αρχές και οι νομικές αρχές θα πρέπει να έχουν καλύτερη ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά τα τρόφιμα στα εθνικά πλαίσια. Να είναι αποτρεπτικά αυτά τα πλαίσια. Δεν πρέπει να υπάρχει κέρδος για τους απαταιώνες ε, από την ε, εξακολούθηση αυτών των ε, δραστηριοτήτων εξαπάτησης. Όλα αυτά πρέπει να διασφαλίζονται στο εθνικό επίπεδο λοιπόν. Καθώς επίσης και οι νομικές σε ε, πράξεις ε, και διώξεις. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις δικές σας όχι ως Προέδρου της Επιτροπής, σας τώρα, αλλά ως σκιώδους εισηγήτριας. Θα ήθελα να πω σημαντικότατα σημεία τα οποία θίγεται, που αφορούν το δίκαιο εμπόριο, περισσότερο αφορούν θέματα εμπορίου με τρίτες χώρες παρά την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό θα ήθελα να εξετάσουν και να δουν οι συνάδελφοι μήπως δεν θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στα θέματα της Επιτροπής μας ε, Ενίας Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν είναι σημαντικά τα θέματα των τροπολογιών σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά δεν εντάσσονται στην επικέντρωσή μας. Ε, εσάς συνάδελφοι σας ευχαριστώ πολύ αλλά και πάλι θα πρέπει να δούμε σε σχέση με τις επιχειρήσεις, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να συνεργαστούμε με τις εταιρείες παραγωγής τροφίμων, αν θέλουμε να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και δεν νομίζω ότι ήταν αποτυχία στην αγορά. Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους ήταν απαταιώνες και εξαπατούσαν Πρέπει όμως να έχουμε όλοι συμφέρον να υπάρχει μια υγιής αλυσίδα, διατροφική αλυσίδα. Διότι όταν κάποιοι ε, κάνουν κάποιες απάτες αυτό υπονομεύει όλους. Γι' αυτό είναι προς όφελος όλων, όλης της κοινότητας ε, που παράγουν, παράγει τρόφιμα να μην υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις απατών. Φοβούμαι ότι δεν είμαι σε θέση πραγματικά να υποστηρίξω την τροπολογία σας, συνάδελφε. Έλαβα υπόψη πλήρως τις τροπολογίες του κυρίου Βίλαντ και του κυρίου Χατζημαρκάκη σε σχέση με τις προτάσεις τους ε, και με τις συμβαστικές τροπολογίες. Και φυσικά προσβλέπω και στις απόψεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσβλέπω στα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω υπό την ιδιότητά μου ως σκιώδους εισηγήτριας. Εξεπλάγιν πρέπει να πω για το ότι κατά το μάλλον ήτον εκπροσωπείται τη θέση ότι όλα βαίνουν λέει καλώς και μόνο θα έπρεπε περισσότερο η εφαρμοσιμότητα και η λειτουργία, ο σεβασμός των νόμων να λειτουργεί. Πραγματικά εδώ δεν ε, το βλέπω να υπάρχει έτσι. Και στο παγκόσμιο εμπόριο έχουμε τρόφιμα τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη και όπου έχουμε ε, απατηλές ε, δηλώσεις, αλλά έχουμε όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και από την παγκόσμια αγορά. Για παράδειγμα, φράουλες στη Γερμανία από την Κίνα. Είναι λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου σημαντικό να πούμε κάποια πράγματα με μια πρόταση ή δύο προτάσεις για την σπουδαιότητα, για την εσωτερική αγορά όλων αυτών αυτών των θεμάτων. Δεν είναι τα πράγματα όπως είπατε εσείς. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κάποια σύντομη παρατήρηση, κάποιο σύντομο σχόλιο γι' αυτό. Λέτε λοιπόν εσείς ότι είναι οι ανώτατες προδιαγραφές που έχουμε εμείς. Στην τροφική όμως αλυσίδα υπάρχουν κάποια κενά, κάποια κάποιες πόρτες και παράθυρα ε, για τους απαταιώνες. Πρέπει να κλείσουμε αυτές τις πόρτες και παράθυρα και δυνατότητες. Και φυσικά αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εθνικά πρέπει να γίνεται. Και όπως σε κάποιες χώρες όπως τη Γερμανία περιφερειακά πρέπει να γίνονται αυτά. Και στην υλοποίηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθούν ως αρρωγή διότι φαίνεται ότι καμιά φορά και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής όλων αυτών κάπως χωλαίνει όταν έχουμε κάποιες ε, επιθεωρήσεις ε, που πριν από ένα μήνα προαναγγέλλονται. Φυσικά οι επιθεωρητές και οι κτηνίατροι που πάνε να κάνουν τέτοιους ελέγχους μόνο εξαιρετικές ε, προϋποθέσεις βρίσκουν στις επιχειρήσεις που πάνε να ελέγξουν. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να γίνονται χωρίς προαναγγελία έλεγχοι και επιθεωρήσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Και φυσικά σήμερα το πρωί πήρα τις συμβαστικές προτάσεις, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, ίσως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες συζητήσεις, να δούμε τι μπορεί να ενταχθεί. Συνολικά, ίσως και για τις τροπολογίες μου, βρίσκω ότι η έκθεσή σας ε, κάπως παρουσιάζει μια αυλαβή, ανώδυνη κατάσταση, εξαπλουστεύει υπερβολικά τα πράγματα και όσον αφορά τα τρόφιμα. Δεν χρειαζόμαστε κάθε δήλωση για κάθε βελόνα που εισάγεται στην Ευρώπη, αλλά για τα τρόφιμα και τα συστατικά τους. Πιστεύω ότι πολιτικοί και οι ε, καταναλωτές χρειάζονται αυστηρότερους κανόνες και αυτό κοστίζει κάτι, είναι δαπανηρό. Γι' αυτό θέσαμε αυτή την τροπολογία να υπάρξει αρρωγή, υποστήριξη που πρέπει να διασφαλίζεται ώστε οι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα μικρά, πολύ μικρά σφαγεία να μπορέσουν να υποστηριχθούν ώστε να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν όλες αυτές οι προτάσεις. Αλλά το ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω κανόνες είμαι πεισμένη γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν η παρέμβαση των σοσιαλδημοκρατών από πλευράς μου ως σκιώδους εισηγήτριας. Τώρα, εδώ για τους πράσινους αλλά πρέπει κυρία Ρούλε είναι σαφές αυτό, να το ξέρουμε ότι είναι από αυτούς. Ο κύριος Χατζημαρκάκης όμως τώρα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να συγχαρώ καταρχήν την εισηγήτρια, συντάκτρια της γνωμοδότησης, διότι από τις 15 τροπολογίες κάνει τρεις συμβιβαστικές με τις οποίες μπορώ να συμφωνήσω γιατί αντικατοπτρίζονται οι απόψεις μου. Δύο-τρεις παρατηρήσεις θα κάνω μόνο. Σχετικά με την πρώτη συμβιβαστική, εδώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας ε, τα οποία θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς μας και τη γραφειοκρατία μας γιατί να το κρύψουμε μπορεί να υπονομεύσει την, τον ανταγωνισμό και την πρόσβαση στην αγορά. Ε, εγώ όμως ε, δεν θέλω πρόσβαση προϊόντων ε, που δεν επιτρέπονται. Οπότε η πρώτη συμβιβαστική σας να είναι ε, όμως α, ενδιαφέρεται οποιαδήποτε νομοθεσία σε αυτό το τομέα, ανησυχεί διότι μπορεί να υπάρξουν λόγω των μέτρων αυξημένες δαπάνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά πρόσβαση στην αγορά για απογορευμένα προϊόντα μην το πούμε. Στη δεύτερη συμβιβαστική, εδώ είμαι ευγνώμων γιατί την τροπολογία μου τη συμπεριλάβατε, δηλαδή την ιδέα μου ότι όλη η τροφική αλυσίδα, αν θέλετε, ε, θα επιτηρείται και ότι θα γίνονται και ευνηδιαστικοί έλεγχοι, αλλά το αποδυναμώνεται λίγο. Λέτε, αναγνωρίζει την σημασία των ευνηδιαστικών ελέγχων. Θα έλεγα ζητή ευνηδιαστικούς ελέγχους. Να το τονίσουμε αυτό και στην τρίτη θα μπορούσε να βελτιωθεί θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτό δηλαδή στην τρίτη συμβιβαστική τροπολογία. Ε, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στην περαιτέρω εργασία σας. Η κυρία Ρουίλε, δυστυχώς τις συμβιβαστικές δεν τις έλαβα. Ε, εγώ ε, δεν μπορούσα να υποβάλω τροπολογίες γιατί είχα άλλη δουλειά. Αλλά θα ζητήσω τμηματικές ψηφοφορίες ίσως είναι σημαντικό να τα ακούσει αυτό η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, τμηματική στην ε, πρώτη για την ε, προαιρετική και το θεσία. Μιλάμε πολύ για αυτήν, αλλά τη θέλουμε και αυτό φαίνεται ε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις για τα τρόφιμα. Όχι θελοντική προαιρετική, αλλά υποχρεωτική ε, σήμανση στα τρόφιμα. Οπότε αυτό το προαιρετική δεν πρέπει να ε, μπει εδώ. Θα ζητήσω τμηματική. Στο σημείο 2, στην τελευταία μισή φράση, ε, έχω αμφιβολίες. Νομίζω ότι πρέπει να διαγραφεί και θα υποβάλω σχετική τροπολογία γιατί περαιτέρω νομικές διατάξεις πρωτίστως είναι προβληματικές γιατί σε ΜΜΕ πιστεύω ότι εκείνοι που δημιουργούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο την τροφική αλυσίδα δεν είναι οι μικρομεσαίες αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν ομήρους τις μικρομεσαίες τη μία ε, απέναντι στην άλλη. Οπότε ε, θα πρέπει να κάνουμε εδώ μια διευκρίνηση ούτω ώστε να ε, είναι πιο σαφές το θέμα για τους καταναλωτές. Για τους μεγάλους ε, παρασκευαστές τροφίμων έχει νόημα να παίρνουν ε, ε, συστατικά από δέκα διαφορετικές χώρες. Αυτό όμως ε, δεν νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Ευχαριστώ. κύριος Μπίλαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Προς την συντάκτρια της νομοδότησης θέλω να πω ότι δεν έχω πολλές παρατηρήσεις, ότι βασικά συμφωνώ με τα όσα παρουσιάστηκαν Συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα και όλα όσα έχουν να κάνουν με την ε, προμήθεια στην διατροφική αλυσίδα. Συμφωνώ επίσης με τις διασυνοριακές κυρώσεις. Όμως έχω κάποιες αμφιβολίες για ορισμένες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε οι αποφάσεις μας να μην αποτελέσουν υπερβολικό άχθος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο σημείο 10 για παράδειγμα. Δεν συμφωνώ ούτε με το σημείο 4, το οποίο ζητάει επιπλέον χρηματοδότηση. Γιατί αναρωτιέμαι πού θα τα βρούμε τα χρήματα αυτά. Τώρα μάλιστα που βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε κι άλλο καλά με την συντάκτρα της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, από την ΚΟΕ e είναι κανείς. Όχι. Και την ομάδα EFD, κύριο Σαβίνη, δεν είναι παρόν. Καλώς. Οπότε κλείνουμε με την εισηγήτρια. Έχετε το λόγο. Και πάλι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι σαφές ε, το γιατί ανέλαβα την έκθεση στην ΙΜΚΟ, γιατί πιστεύω ότι είναι κέριο θέμα των καταναλωτών και ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε και τη δυνατότητα πρόληψης και, τη δυνατότητα δίωξη, δίωξης της απάτης. Οπότε δεν δέχομαι την επίθεση από πράσινους και κόκκινους ότι απλουστεύουμε τα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι καλά τα πράγματα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό που λέω είναι ότι ούτε, ε, ούτε, η κυρία Ρούλε, ούτε εσείς δώσατε συγκεκριμένες προτάσεις. Πείτε μας συγκεκριμένα ποιοι νέοι κανόνες, μέσα από ποια νομοθεσία, ποιος θα πληρώσει το κόστος, πού είναι η προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές. Όταν υποβάλλετε τροπολογίες τέτοιες, τότε θα βάλω θετικό πρόσημο στην, στον κατάλογο της ψηφοφορία. Τώρα όμως έχουμε μόνο παράπονα, ε, αλλά... Ε, αν δεν υπάρχουν, ε, δεν προωθούνται τα θέματα, δεν φταίω εγώ, τα δικά σας. Ε, για τα κενά τώρα, για τα παραθυράκια. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να συνεργαστούμε με Προεδρία και κράτη-μέλη για να φροντίσουμε ότι θα λάβουν εκείνη μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να ενισχύσουν τις κυρώσεις, τα πρόστιμα, τους ελέγχους. Εγώ έκανα μια τροπολογία με συναδέλφους για να ζητήσω ευνηδιαστικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις. Και Μπορώ να το αλλάξω. Όχι αναγνωρίζει, να αποζητεί. Βεβαίω συμφωνώ μαζί σα, Είναι η τροπολογία μου. Διαβάστε τη. Επίσης, κυρία Πρόεδρε, ε, σα ρωτώ σκιώδη, όταν λέτε ότι πρέπει να δώσουμε χρήματα και ενισχύσει μεσούσεις της χειρότερης χρηματοπιστωτικής κρίσης σε, στην Ευρώπη και στον κόσμο σε ΜΜΕ ε, που είναι η πλειοψηφία στην ε, τροφική ελισίδα η οικονομική κάλυψη ποια θα είναι, ποιος θα πληρώσει, ποιες μικρομεσαίες θα λάβουν χρήματα, ποιες όχι, ποια τεράστια γραφειοκρατία και σε ποιο επίπεδο θα δημιουργήσετε για να διαχειριστούν τα χρήματα. Κάντε προτάσεις που θα είναι εφαρμόσιμες στην πραγματική ζωή. Μην κάνετε ρητορίες και ανακοινώσεις επιθεμάτων που δεν υλοποιούνται και δεν δίνουν και προστιθέμενη αξία στους παταναλωτές. Γι' αυτό βάζω αρνητικό πρόσημο και λέω ότι πρέπει να ενισχύσουμε η αδίποτε εταιρεία τροφίμων στην Ευρώπη για το κόστος των πρόσθετων ε, επιθεωρήσεων. Καλύτερα να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα επιθεωρήσεων που δεν θα δημιουργεί γραφειοκρατία ούτε πρόσθετες δαπάνες για τις μικρομεσαίες και τους καταναλωτές. Θα αποτρέπει όμως ε, τις απάτες με τα τρόφιμα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και νομίζω ότι συμφωνούμε στην ανάλυση αυτή. Απλώς υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόβλημα με οτιδήποτε έχει σχέση με αυτορυθμίσεις και συνεργασία με τον κλάδο. Θέλετε να τιμωρήσετε τη βιομηχανία. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει τους καταναλωτές. Σίγουρα λαμβάνω υπόψη τα δύο σχόλιά σας, κύριε Χατζημαρκάκη, και θα κάνω τις σχετικές τροποποιήσεις Τέλος να πω ναι για την λασιμότητα. Όταν έχουμε συνεργαστεί στη συνεργασία ετικετοθεσίας, εγώ υπέβαλα τροπολογίες όταν είχαμε συνεργαστεί δηλαδή για την ε, ετικετοθεσία είχα κάνει τροπολογίες ούτω ώστε να υπάρχει ε, σήμανση προέλευσης όλων των κρεάτων. Και νομίζω ότι ο καταναλωτής δικαιούται να ξέρει την προέλευση του κρέατος, να αυξήσουμε την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια δηλαδή. Αυτό που λέω και το επαναλαμβάνω εδώ γιατί βλέπω την πραγματικότητα των μικρομεσαίων, έχω και εγώ, μην το κάνουμε όμως με τρόπο που δεν εφαρμόζεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε καταγωγή όλων των ε, συστατικών των τροφίμων ε, σε κάθε τρόφιμο που έχει 1,1, 0,1 ε, κρέας. Συμφωνώ όμως με τι κυρίε Ρούλε και Βάιλερ ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ίχνη λασιμότητα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, τελειώνω εδώ και θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη μου όσο γίνεται περισσότερα από τα θέματα που θέσατε και την τελευταία παρατήρηση στη συμβιβαστική τροπολογία και κυρίες Ρούλε και Βάιλερ, αν θέλετε να συνεχίσω με το διάλογό μας, πάντα είμαι πρόθυμη για κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια. Είναι αυτονόητο ότι τώρα δεν θα επισέθω σε περισσότερες λεπτομέρειες θα συζητηθούν αυτά και μια και ο πρόεδρος μας δεν παρίσταται ακόμα, δεν έχει ακόμα επιστρέψει και έχει αυτές τις συζητήσεις με την Βρετανική κυβέρνηση, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, μικρό διάλειμμα, τεσσάρων λεπτών ίσως, όπου επίσημα θα περάσουμε μετά στις ψηφοφορίες. make Okay. Uh, so, uh, ladies and gentlemen, Κυρίες και κύριοι, ας αρχίσουμε τις προφορίες μας, παρακαλώ. Σας παρακαλώ όλους να καθίσετε πρώτα απ' όλα. Έχουμε διάφορες σημαντικές ψηφοφορίες σήμερα. Θα ψηφίσουμε και ηλεκτρονικά, έτσι, όπως κάνουμε συνήθως, οπότε ελπίζω να έχετε τις κάρτες σας. κύριε Κέπαρτ και ο κύριος Σβάμπ ή ποιος, κύριε Χάνσλεϊ, ναι, εκείνη που θα ηγηθεί και θα για να ξέρω ποιοι θα δείχνουν ε, τι ψηφίζουν οι ομάδες, για να ξέρω αν πρέπει να περνάμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία ή όχι. Ωραία, έτσι το ξέρω τώρα. Λοιπόν, πάλι παίρνω το αριστερό μικρόφωνο γιατί έτσι φαίνομαι καλύτερα στο web stream, λέει ο πρόεδρος. Πρώτο σημείο λοιπόν στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ ησυχία. Ας ακούσουμε πρώτα την εισηγήτριά μας, την κυρία Βάιλερ, η οποία ζητάει εντολή για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου όσον αφορά τον ραδιοεξοπλισμό. Νομίζω ότι η ψήφος στην Επιτροπή για αυτή την οδηγία ήταν τόσο σαφής χωρίς ε, αρνητικές ψήφους, χωρίς αποχές, όλοι ψήφισαν υπέρ, ώστε μπορούμε με εμπιστοσύνη να πάμε στον τριμερή διάλογο εάν συμφωνήσει σήμερα η Επιτροπή. Θα ήμουν ευγνώμων και όλοι οι σκιώδεις με τους οποίους έκανα τη Δευτέρα μια, μια πρώτη συζήτηση επ' αυτού μου είπαν ότι και εκείνοι συμφωνούν, οπότε έχουμε μια ευρία βάση από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Θα δείτε ίσως ότι στην απόφαση, δεν ξέρω αν υπάρχει, πάντως στην απόφαση έχουμε προσθέσει ότι περιμένουμε από το Συμβούλιο να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα γιατί οι συζητήσεις ήταν λίγο κατακαιρματισμένες με το Συμβούλιο και θα είναι δύσκολο ε, να καταλήξει σε κοινή θέση το Συμβούλιο. Γι' αυτό συμφωνήσαμε να έχουμε μία προθεσμία μέχρι 20 Δεκεμβρίου για τις διαπραγματεύσεις, ώστε να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κοινή θέση. Αν δεν υπάρξει, τότε στις αρχές του έτους θα σκεφτούμε ποια νέα βήματα θα κάνουμε. Καταρχήν όμως έχουμε εμπιστοσύνη και είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να αρχίσουμε τον τριμερή διάλογο. Και ε, παρακαλώ όλους τους συναδέλφους, τις συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ. Ωραία, θα ψηφίσουμε για να έχετε την εντολή και σας ευχαριστούμε για το μέχρι τώρα έργο σας. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Με 38 οι κάρτες μέσα, αλλά 33 ψηφίζουν. Πέρα τη ψηφοφορία. Η κυρία Ταμπέλα δεν έχει την κάρτα της. 33 υπέρ και μία ψήφος κατά. Ωραία, η εντολή είναι σαφής γιατί χρειάζονται πάνω από τα μισά μέλη της Επιτροπής μας, υπάρχουν. Είσαστε υπέρ ή κατά εσείς. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι σαφές. Χρειαζόμαστε πάνω από τα μισά μέλη της Επιτροπής που τα έχουμε. Οπότε καλή τύχη κύριε Βάιλερ. Επιβεβαιώνω ποια είναι η διαπραγματευτική ομάδα. Εγώ ως πρόεδρος, η κυρία Βάιλερ ως Μάτι Κέιν, Μάντες, Ρούλε και Σαβίνη. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στην γνωμοδότησή μας προς την ε, Επιτροπή Εμπορίου για την πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ο κύριος Έγγελ είναι ο εισηγητής μας. Δεν τον βλέπω όμως εδώ. Οπότε περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Τροπολογίε 15 και 16 που είναι ίδιες για απόρριψη της πρόταση. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Μια στιγμή. Ξανά. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Οπότε, περνάμε στην υπόλοιπη ψηφοφορία. Έχουμε μια μπλοκ ψηφοφορία, ένα, όλες μαζί, βλέπετε ποιες είναι, υπέρ, κατά εγκρίνονται. Οπότε περνάμε τώρα στην τροπολογία 47. Υπέρ παρακαλώ. Α, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 47. 41 κάρτες είναι στο μηχάνημα. Ψηφίστε πιο γρήγορα. Αν θέλετε να ψηφίσετε, ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 22 κατά 18 υπέρ. Α, 19. Έχετε την κάρτα εσείς δεν την έχετε μαζί. Καλά, θα υπολογίζω και την ψήφο σας. Λοιπόν, τροπολογία 48 τώρα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Η κυρία Σβέλλα είναι υπέρ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 22 ψήφοι υπέρ 18 κατά. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 50 και τις επόμενες που θα ψηφίσουμε όλες μαζί. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνονται. Τώρα. 51 του κυρίου Ταραμπέλα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 51. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτεται. 16 υπέρ, 25 κατά. Συμβαστική τροπολογία αριθμός 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πατάτε το κουμπί όσο γίνεται πιο γρήγορα παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Αφού απορρίφθηκε 54. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57 καταπίπτει. 58 τώρα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 58. Πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα πάλι σε... Α, στην 65 πρώτα, συγγνώμη ο πρόεδρος του κυρίου Λόκεκα. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τώρα περνάμε σε μια σειρά τροπολογιών. Block vote 3. Υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 67 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε καλύτερα για την 88. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της προφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 90 τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 91. Ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 96 καταπίπτει. Σωστά. Ναι. 99 λοιπόν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για την τροπολογία 100. Ψηφίστε. Πέρα τη υποφορίες, απορρίφθηκε. Τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 10. Του συγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 106. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11 του Σιγητήπερ. υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 107. Ψηφίζουμε. Είναι 107 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάλι τώρα μαζικά ψηφοφορίες μπλοκ 4. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 112. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 116 και 117 μαζί. Υπέρ. Κατά απορρίπτονται 118 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 119 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 120 ε, αυτή καταπίπτει. Όχι, 120 την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 12 και 13 μαζί υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 14 του συγκεκριτή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά, 126 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 125 καταπίπτει, 124 ως προσθήκη. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται η προσθήκη. Ερχόμαστε τώρα στα αιτιολογικά. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 18 ως προσθήκη, Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ομαδοποιημένα τώρα, ε, η 7, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 21, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 19, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 22, όχι. 22 συνολικά υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 33 και 35 μαζί, υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 37 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 40 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα ηλεκτρονικά. Είναι 43 μέλη παρόντα. Είναι ένας παραπάνω. Ας βάλει κάποιος την κάρτα. Ένας από τους σοσιαλιστές παραπάνω είναι. Οπότε κάποιος από τους σοσιαλιστές... Α, ε, εσείς την έχετε την κάρτα σας μένα, αλλά βγάλτε την, γιατί αφού είναι ένας παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Συνεπώς, 28 ψήφοι περ, 11 κατά και καμία αποχή. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Έγγελ. Κύριε Βάιλερ, θέλετε να πείτε κάτι, παρακαλώ. Η κυρία Βάιλερ εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών, αγαπητοί συνάδελφοι, διακόπτει η ομιλήτρια. Θα ήθελα τουλάχιστον μια σύντομη παρατήρηση να κάνω στη συνολική αυτή διαδικασία. Χθες το βράδυ, γύρω στις 10 το βράδυ, από πλευρά του έμαθα γιατί όλες τις δικές μας σοσιαδημοκρατικές τροπολογίες τις απορρίπτει. Και θέλω να πω δεν είναι δίκαιο και αλληλέγγυο από πλευρά συμπεριφοράς σε συναδέλφους αυτό. Και πρέπει να μας εξηγήσει γιατί ήταν εναντίον. Το βρίσκω θλιβερό ότι σε ένα τόσο σημαντικό χαρτοφυλάκιο που έχει σημαντικές επιπτώσεις και συνέπειες και που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και συνέπειες για την παγκόσμια πολιτική εμπορίου όλες τις δικές μας τροπολογίες, σχεδόν όλες από τις 28 τροπολογίες τις απέρριψε. Η πρόταση της Επιτροπής θα έπρεπε να μπορούσε να έχει βελτιωθεί με αυτές τις τροπολογίες μας και απουσιάζει η κοινωνική ισορροπία όσον αφορά την ισορροπία των κοινωνικών ε, θεμάτων και συντελεστών. Και για το αντίστοιχο άρθρο που εμείς πιστεύουμε ότι το σύνολο αυτό των προτάσεων θα μπορούσε να, είχε, να, θα μπορούσε να ε, γίνει δεκτό, είναι σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα ότι οι όροι και προϋποθέσεις στην παγκόσμια αγορά θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε για τους παγκόσμια εμπλεκόμενους global players να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλω όμως να πω ότι τη διαδικασία αυτή από πλευρά εισηγητού δεν την θεωρώ αλληλέγγυα και φιλική προς συναδέλφους ως ήθιστε να ακολουθείτε ε, στο Ευρωκοινοβούλιο και στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, λοιπόν, εντάξει, ο πρόεδρος όμως δεν μπορεί <clears throat> να διευθετήσει ή να επιβάλλει κάποιες απόψεις σε τέτοια θέματα. Υπήρξε νομίζω ευκαιρία για τη συζήτηση αυτών των τροπολογιών, συζήτηση των τροπολογιών στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και από πλευράς χρονοδιαγράμματος υπάρχει χρόνος ώστε να συζητώνται αυτά τα θέματα δημόσια και ανοιχτά. Όμως οι συνάδελφοι πολλές φορές όταν δεν παρίστανται για αυτές τις συζητήσεις Δυσχεραίνουν τα πράγματα. Εσείς κυρία θέλετε να ομιλήσετε εξ ονόματος του εισηγητού. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σήμερα, εδώ εκπροσωπώ τον εισηγητή. Από ό,τι γνωρίζω, ο εισηγητή ακολούθησε την εξή στάση. Στην συνεδρίασή μα είχαμε χρόνο να συζητήσουμε για όλε αυτέ τι τροπολογίε. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει χρόνος να ανταλλάσσουμε απόψεις. Λοιπόν, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανονισμοί και οι κανόνες και έτσι να εργαζόμαστε. Ενθαρρύνουμε όμως και υποστηρίζουμε οι συγητές να συναντώνται σε τακτά διαστήματα με τους κοιόδης συγητές ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το έργο τους. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στην ώρα να ψηφίσουμε την έκθεση Σάντεμος για την πρόταση για ένα κανονισμό για την ασφάλεια προϊόντων όσον αφορά τους καταναλωτές. Μια πρόταση που επί μεγάλο χρονικό διάστημα εργαζόμαστε επ' αυτής στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο Ελπίζω ότι μπορεί να θα μπορέσει να σημειωθεί πρόοδος ε, με στόχο να μπορέσουμε <clears throat> να ε, ολοκληρώσουμε το έργο μας ε, έγκαιρα και με την έγκριση των συντονιστών να υπάρχει και αρκετός χρόνος για την διαπραγμάτευση όλων αυτών. Προτού περάσουμε στην ψήφιση, κάποιος εισηγητής ή άλλος θέλει να κάνει παρατηρήσεις ή περνάμε αμέσως στην ψήφιση. Κυρία Σαντεμόζε παρακαλώ. Συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλά και μόνο να πω το εξής. Έχουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε, πιστεύω, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο πριν από την εκπνοή αυτής της κοινοβουλευτικής εντολής. Να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, λοιπόν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν συμφωνήσει, συμφωνούν επ' αυτού. Α ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Δεύτερον, μια παρατήρηση για τον πίνακα ψηφοφορία. Κατά τις τελευταίες 24 ώρες, πολύ πρόσφατα, υπήρξαν κάποια προβλήματα ίσως σε σχέση με τον πίνακα αυτόν. Μια ασυνήθιστη, ας το πω έτσι, διαδικασία και απογοητεύτηκα γιατί ουσιαστικά δεν είχα εμπλακεί και θα έπρεπε να είχα εμπλακεί ως εισηγήτρια σε όλα αυτά. Τώρα όμως έχουμε ένα πίνακα ψηφοφορίας που συντάχθηκε, εν πάση περιπτώσει και μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά Θέλω να το πω και να εισακουστεί ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο καταλήξαμε και εργαστήκαμε για αυτόν την πίνακα ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου για τι συζητήσει για τον κανονισμό για την ασφάλεια προϊόντων για του καταναλωτέ. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μπαλτασάρε για μια πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Και στο τέλος τέλος οι καταναλωτές νομίζω θα ε, επωφεληθούν και θα πρέπει να ευχαριστούν το Κοινοβούλιο για τα ε, θετικά αποτελέσματα. Ας προχωρήσουμε στην ψήφιση λοιπόν. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Κύριε Παντασάρ, εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να το θίξω και να το αναφέρω αυτό, αυτό το οποίο ανέφερε προηγούμενα η συγγήτρια. Χθε είχαμε μια προφορική τροπολογία που ε, παρουσιάστηκε, προφορική τροποποίηση που προτάθηκε. Η συγγήτρια όμως ε, δεν ήθελε, δεν συμφωνούσε. Στις 7 η ώρα καταλήξαμε σε ε, μια συμβαστική τροπολογία από αυτή την πρόταση, αρχική πρόταση. Ίσως είναι δυσάρεστο αυτό το οποίο έγινε τελικά, αλλά όμως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα για την έκθεση, ώστε στις 20.00 ε, στις 8 η ώρα το βράδυ να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Όμως παρόλα αυτά πιστεύω ότι η γραμματεία, το άρθρο 161 του κανονισμού, ε, που ήθελε να εφαρμοστεί, δηλαδή ότι υφίσταται η δυνατότητα και μετά τη συζήτηση να υπάρξει μια συμβαστική τροπολογία που θα, μπορεί, μπορούσε να κατατεθεί. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται όμως επιπλέον ότι το Κοινοβούλιο για τέτοιου είδους ε, συμβαστικές τροπολογίες, την τροπολογία 10, θα μπορούσε να ψηφίσει. Όμως εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή η συμβαστική τροπολογία θα μπορούσε να γίνει δεκτή και θα έπρεπε να εγγραφεί στον κατάλογο ψηφοφορίας. Και όσον αφορά τη μεθοδολογία, νομίζω δεν είναι η σωστή μεθοδολογία και η σωστή προσέγγιση. Δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εργαζόμαστε στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, το συζητήσαμε αυτό στους συντονιστές ε, στη συνάντηση συντονιστών σήμερα το πρωί, κύριε Μπαντασάρη. Η κυρία Σάντε Μόζε είπε ότι παρότι κατατέθηκε αργά αυτό, αυτός ο συμβιβασμός και είχε ε, υποβληθεί από δύο κοινοβουλευτικέ ομάδες. Γι' αυτό είναι αποδεκτός και μπορεί να ενταχθεί στον πίνακα ψηφοφορίας. Δεν έχω άλλη δυνατότητα παρά να ψηφίσουμε. Αν εσείς δεν θέλετε μπορείτε να καταψηφίσετε. Αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Αν ήταν κατά των κανόνων δεν θα το είχα δεχτεί, δεν θα είχε ενταχθεί στον πίνακα ψηφοφορίας με κάποια παρατήρηση ότι υπήρξε καθυστέρηση συμφωνώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα διευθετηθεί ψηφίζοντας. Αν απορριφθεί έληξε. Γι' αυτό λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καταλήξαμε σε αυτό το συμβιβασμό που εντάχθηκε ώστε να μπορεί να υπερψηφιστεί, να καταψηφιστεί αν δεν επιθυμείτε. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κάνουμε λόγο για τον συμβιβασμό 10, αυτός είναι ο συμβιβασμός περί του οποίου ο λόγος. Μάλιστα, ως, ε, ελάχιστο, ως ελάχιστη προϋπόθεση θα μπορούσε από δύο κοινοβουλευτικές ομάδες να κατατεθεί. Λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα και προφορικές τροποποιήσεις να τις απορρίπτετε. Εφόσον λοιπόν κάποιοι διαφωνούν, δεν θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές τέτοιες προφορικές τροποποιήσεις. Προχωράμε. Βιομηχανική, ε, Επιτροπή Βιομηχανίας 1. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 112. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 35 της εισηγήτριας υπέρ, κατά εγκρίθηκε. Γι' αυτό περνάμε αμέσως στην γιούρη 4, νομικών υποθέσεων 4, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 5α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Διεθνούς εμπορίου 11, υπέρ, κατά, Φύσουμε ηλεκτρονικά για να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία Είναι τα 11. Άρχεται. Να επιταχύνετε παρακαλώ την ψήφιση. Έχουμε 34 κάρτες που έχουν δικαίωμα ψηφίσουν, 39 όμως συμμετέχουν. Εγκρίθηκε 21 υπέρ 18 εναντίον. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό και υπάρχουν κάποιοι παραπάνω με τις κάρτες, αλλά εν πάση περιπτώσει. εντάξει, συμβαστική τροπολογία 7α υπέρ κατά, εγκρίθηκε, είναι σαφές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 117 υπέρ, υπέρ. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Πρέπει να πάμε στο συμβασμό 1 πρώτα. Συμβαστική τροπολογία 1. Δημιουργήθηκε μια σύγχυση, ζητώ συγγνώμη. Συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά. Σαφώς εγκρίθηκε. Τροπολογία 117 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Ήτρε 18 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 118 υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας καταψηφίστηκε Τροπολογία 119 υπέρ. Υπέρ και πάλι 119 κατά. Απορρίφθηκε, είναι σαφές το αποτέλεσμα. Τροπολογία 120 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 122 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε νομικών υποθέσεων Γιούρι 5 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Είναι τα 12 και τροπολογία 123 από κοινού υπέρ αυτών υπέρ υπέρ κατά εγκρίθηκαν, είναι σαφές το αποτέλεσμα, εγκρίθηκαν. Τροπολογία 121 υπέρ 121 κατά Α, θα Ο ΜΟΥ μάλιστα. Εντάξει. Είναι μέρος της συνολικής ψηφοφορίας. Ήταν στο σύνολο των τροπολογιών. Η έγκριση, η... το αποτέλεσμα είναι για το σύνολο αυτών. Τροπολογία συμβαστική 6α υπέρ κατά. Σαφώς εγκρίθηκε. 125 τροπολογία υπέρ Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε την τροπολογία 125. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 38 καταπίπτει. 38. Ήτρε 20. Επιτροπή Βιομηχανίας 20. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 128 καταπίπτει. Ήτρε Βιομηχανίας 21. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Παρακαλώ, συγγνώμη. Κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 129 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 130 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 131 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 39 και 134 υπέρ αυτών κατά απορρίφθηκαν αυτές οι δύο. Τροπολογία 132 και 136 από κοινού υπέρ κατά εγκρίθηκαν. 133 καταπίπτει 135 καταπίπτει, 140 καταπίπτει, πάμε στην 137 υπέρ. Κα, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 138 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Η τρέβιο 22 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 139 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 141 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 40 με και προφορική τροποποίηση, με προφορική τροποποίηση που υποθέτω γίνεται δεκτή από την εισηγήτρια. Υπέρ αυτής κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 41 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 142 αποσύρθηκε. Η 13 διεθνούς εμπορίου υπέρ κατά απορρίφθηκε. Βιομηχανίας 23 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 42 με προφορική τροποποίηση της ΑΡΔΕ που εμφαίνεται από τον πίνακα ψηφοφορίας. Μπορούμε όλα αυτά να τα πάρουμε με την προφορική τροποποίηση. 42 με προφορική τροποποίηση. Εντάξει, υπέρ αυτής. Κατά εγκρίθηκε. Ήτρε, βιομηχανίες 24, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 143 τροπολογία, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 144, καταπίπτει, μάλιστα, καταπίπτει 144. Και βιομηχανίας 25 καταπίπτει επειδή είχαμε συμβιβασμό. Και πάμε τώρα στην 145 και ψηφίζουμε με προφορική τροποποίηση που διαγράφει το or, το e. Τι θα κάνουμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν με την προφορική τροποποίηση. Ωραία, είναι αναπόσπαστο μέρος. Υπέρ λοιπόν, κατά, απορρίφθηκε. 146 καταπίπτει και πάμε στην 147 υπέρ. Κατά, απο, α, απορρίφθηκε. 148 καταπίπτει. 149 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Η 43 υπέρ κατά απορρίφθηκε η 43. Η 151 υπέρ κατά και αυτή απορρίφθηκε. Η 150 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Είναι τα 14 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 153. Καταπίπτει αυτή. Επειδή εγκρίθηκε ο συμβασμός 7β, αποσύρθηκε η 45. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο προς τον πρόεδρο δεν ακούστηκε. Η τροπολογία 155 υπέρ κατά απορρίφθηκε 156 υπέρ κατά απορρίφθηκε 158 και είναι τα 15 υπέρ αυτών κατά εγκρίθηκαν βιομηχανίας 28 υπέρ κατά απορρίφθηκε βιομηχανίας 29 υπέρ κατά απορρίφθηκε οι 159 και οι 160 υπέρ αυτών. Νομίζω πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 159 και 160 ψηφίζουμε. Άρχεται. Ομού και οι δύο. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν αυτές οι δύο τροπολογίες. Συμβιβασμός, συμβιβασμός 7β υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Είναι σαφές το αποτέλεσμα η 143 κατέπεσε για τα πρακτικά. Και πάμε τώρα στην συμβαστική 2α υπέρ κατά εγκρίθηκε. Και πάμε στην τροπολογία 167 υπέρ απορρίφθηκε. 168 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 154 καταπίπτει γιατί εγκρίναμε το συμβασμό 7β ή 169 τώρα υπέρ κατά απορρίφθηκε η 171 και η 172 και η 31 υπέρ αυτών των τριών κατά εγκρίθηκαν οι τρεις τροπολογίες. Γιούρι 8 υπέρ κατά απορρίφθηκε Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε αυτή την τροπολογία ηλεκτρονικά. Θα ελέγξουμε για να βεβαιωθούμε ότι όλοι γνωρίζουν το τι συμβαίνει. Λοιπόν, ψηφίζουμε την Γιούρι 8, την νομικών υποθέσεων τροπολογία 8, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν η τροπολογία αυτή με τρεις ψήφους διαφορά, 21 υπέρ 18 εναντίον, η 48 καταπίπτει, η 173 τώρα υπέρ κατά απορρίφθηκε, είναι σαφές το αποτέλεσμα. Οι 49 και 174 αποσύρθηκαν, οι 175 τώρα με προφορική τροποποίηση που νομίζω η συγγήτρια την δέχεται. Υπέρ αυτής, κατά, εγκρίθηκε. Οι 176 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Οι 177 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Η 50 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 51 τώρα. Και σύνολο ψηφοφορίας μαζί με αυτήν υπέρ, κατά, αυτή η ομάδα εγκρίθηκε. Η 180 τώρα υπέρ, κατά, απορρίφθηκε η 180. 181 και βιομηχανίες 33 υπέρ αυτών των δύο, κατά, εγκρίθηκαν. Η 170 καταπίπτει. Είναι τα 16 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Η 152 καταπίπτει και πάμε τώρα στον συμβιβασμό 4, συμβιβαστική 4, εντάξει, συμβαστική 4, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Πάμε τώρα, ένα σύνολο τροπολογιών έχουμε στο άρθρο 7, υπέρ αυτών, κατά, απορρίφθηκαν, είναι σαφές. Πάμε στο άρθρο 7. Θα ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε. Είναι για διαγραφή αυτή η τροπολογία. Έτσι. Είναι υπερδιαγραφή του άρθρου 7. Για να είναι σαφές το τι κάνουμε. Διαγράφεται όλη η παράγραφος. Και μετά θα ψηφίσουμε τη συμβαστική 10. Τροποποιημένη διατύπωση του άρθρου 7. Και αν καταπέσει και αυτό θα ψηφίσουμε τις επόμενες. Δηλαδή στόχος είναι αυτών των τροπολογιών να διαγραφεί το άρθρο 7. Άρχεται η ψήφιση όλων αυτών των τροπολογιών για διαγραφή. Είναι σημαντικό να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Πέρας ψηφοφορίας επ' αυτών. Απορρίφθηκαν, είναι σαφές. Οπότε απορρίφθηκαν οι τροπολογίες για διαγραφή. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά στη συμβιβαστική 10. και μετά θα ψηφίσουμε καθένα από τα άρθρα όπως ε, προβλέπετε στην αρχική διατύπωση. Πέρας ψηφοφορίας. Η συμβαστική τροπολογία 10 απορρίφθηκε, είναι σαφές. Και περνάμε τώρα και ψηφίζουμε τις επιμέρους τροπολογίες ε, ως ακολουθούν, όπως ακολουθούν. Αρχίζουμε με την International Trade Διεθνούς Εμπορίου 17 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε η 17 του Διεθνούς Εμπορίου. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Να ελέγξουμε λέγεται στον Πρόεδρο. Είσαστε εναντίον εσείς. Ωραία. Η 17 του Διεθνούς Εμπορίου. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Να ψηφίζετε πιο γρήγορα παρακαλώ συμμετέχοντα στην ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορία τώρα. Και απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Τώρα, 192, τροπολογία 192. Όσοι είναι υπέρ, κατά, Απορρίφθηκε, είναι σαφές. Η 191 τώρα, υπέρ. Κατά. Α, να το ελέγξουμε. Η 191. Ψηφίζουμε την 191, άρχεται η ψηφοφορία. Για να είμαστε βέβαιοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και σαφώς απορρίφθηκε η 191. Γιούρι 10. Υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 193 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 195 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 194 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Ίντα 18 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Ίντα 19 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Είναι τα 20 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 196 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Είναι τα 21 υπέρ υπέρ κατά απορρίφθηκε. Είναι σαφές. Η τροπολογία 197 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Η 198 υπέρ κατά απορρίφθηκε 199 υπέρ κατά εγκρίθηκε η 199 και έτσι τώρα ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες για το άρθρο 7 και περνάμε στο άρθρο 8 συμβιβασμός 8α σε τμήματα ψήφιση όπως ζητήθηκε από την ομάδα ALDE αυτό που θα κάνουμε είναι θα ψηφίσουμε τα διαφορετικά τμήματα αυτής της συμβαστικής τροπολογίας. Πρώτα το πρώτο τμήμα υπέρ του πρώτου τμήματος και συμβαστικής τροπολογίας 8. Υπέρ κατά σαφώς εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα υπέρ κατά και το δεύτερο τμήμα εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε το άρθρο το τρίτο τμήμα. Τρίτο τμήμα της 8 συνεχίζεται και συνεχίζεται η ξεχωριστή ψήφιση με το αίτημα τσάντε. Σε τμήμα λοιπόν ψηφοφορία για το 3 υπέρ κατά εγκρίθηκε το τρίτο τμήμα και μετά έχουμε μια προφορική τροποποίηση που νομίζω γίνεται δεκτή από όλους, έτσι, η προφορική τροποποίηση, υπέρ λοιπόν αυτής. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα, για την έκβαση είναι τμήμα λοιπόν τη συμβαστική τροπολογία η προφορική αυτή τροποποίηση με αυτόν τον τρόπο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία και αποτέλεσμα ισοψηφία. Απορρίφθηκε 19-19. Και νομίζω υπάρχει και ένα τελικό τμήμα αυτής της προφορικής ε, τροποποίησης που ζητήθηκε Σωστό. Μια δεύτερη προφορική τροποποίηση που αντικαθιστά το must με το should. Όσοι είναι υπέρ λοιπόν, υπέρ της αντικατάστασης, κατά τώρα. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Να αρχίσουμε να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αποτέλεσμα εγκρίθηκε με μια ψηφοδιαφορά 19 υπέρ 18 εναντίον. Εντάξει. Και τώρα, σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, περνάμε κατευθείαν στη συνέχεια. Πού πάμε ακριβώς τώρα, σε ποια τροπολογία. Έχουμε διάφορε, διάφορες σελίδες παρακάτω που συνεχίζουμε. Τροπολογία 255 κυρίου Φόξ. 255, συμφωνείτε, αυτή θα ψηφίσουμε. 255 του κυρίου Φόξ. Όσοι είναι υπέρ της 255. Κατά εγκρίθηκε η 255. Και τώρα έχουμε τον συμβιβασμό 8β υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Και πάμε στη συνέχεια στη συμβιβαστική τροπολογία 8γ, 8c. Ε, Κάποιες σελίδες παρακάτω και αυτή. Και πάλι έχουμε σε τμήματα ψήφιση που ζητήθηκε από την Άλντα εδώ είναι υπέρ των ξεχωριστών ψηφοφοριών οι άλτε σήμερα. Πρώτο τμήμα λοιπόν της 8 γ χωρίς την παράγραφο 4α υπέρ. Κατά εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά και αυτό το δεύτερο τμήμα εγκρίθηκε. Και περνάμε στην συνέχεια στην τροπολογία 303. Αποσύρθηκε αυτή. 304 του κυρίου Σαλβίνη υπέρ της 304. Κατά Απορρίφθηκε η 304. Τροπολογία 305 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 306 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 307 υπέρ. υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Συμβαστική τροπολογία 9. Σε τμήματα ψήφιση ζητήθηκε από την εισηγήτρια. Σωστό. Μάλιστα. Όχι. Εντάξει, αυτό τουλάχιστον σύμφωνα με τον δικό μου πίνακα ψηφοφορία. Το σύνολο θα ψηφίσουμε, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Υπέρ τη 9. Συνολικά. Κατά. Η 9 εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 9 εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 322. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 3 324 υπέρ κατά απορρίφθηκε η 324 323 υπέρ κατά απορρίφθηκε 326 υπέρ κατά απορρίφθηκε 325 υπέρ κατά απορρίφθηκε 328 υπέρ κατά απορρίφθηκε 327 υπέρ κατά απορρίφθηκε 329 και 51 υπέρ αυτών υπέρ κατά εγκρίθηκαν οι 330 υπέρ κατά απορρίφθηκε Ήτρε 52 υπέρ κατά απορρίφθηκε τροπολογία 64 υπέρ κατά απορρίφθηκε τοπολογία 67 Η 67 λοιπόν υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 331 και ήτρε 53 υπέρ αυτών. Κατά. Εγκρίθηκαν. Τροπολογία 332 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Ήτρε 54 υπέρ. Υπέρ Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να δούμε τι γίνεται. Ασαφές ήταν το αποτέλεσμα. Ήτρε 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Με δύο ψήφους διαφορά μόνο. Έστω. Τροπολογία 333. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Ήτρε 55. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τοπολογία 334 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Γιούρι 15 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 335 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τοπολογία 336 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε η 336. Και η 56 τώρα, υπέρ. Υπέρ. Δεν βλέπω κανείς να είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Mm. Από το ΕΛΚ. Ωραία, έστω. Η 56 είπαμε. Η 356. 56. Εντάξει. Λοιπόν, Είμαστε στην Ήτρε 56 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 65 τώρα. Της κυρίας Αλντεμόζε υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Είναι σαφές. Τροπολογία 337 και Ήτρε 57 υπέρ αυτών. Κατά. Εγκρίθηκαν. Τροπολογία 338 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Ήτρε 58 υπέρ κατά να απορρίφθηκε η 69 υπέρ απορρίφθηκε τροπολογία 70 της εισηγήτριας υπέρ κατά απορρίφθηκε συμβιβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά εγκρίθηκε Πάμε στην τροπολογία 352, ε, Γιούρι 16, Γιούρι 16 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε, είναι σαφές. Ε, ήτρε 60 υπέρ, υπέρ της Ήτρε 60, κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Της Επιτροπής Βιομηχανίας τροπολογία 16, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά επ' αυτής. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 19-19 ισοψηφία καταψηφίστηκε. Ευτυχώς το ελέγξαμε. Περνάμε τώρα στην Επιτροπή Βιομηχανίας 61. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 73 καταπίπτει. 74 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε η 74. 75 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Μπορούμε ομού να ψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες. Της εισηγήτριας. Συμφωνείτε. Με, από το 1 έως το 6 τροπολογίες. 1 έως 6 λοιπόν ομού. Όχι, δεν συμφωνείτε εσείς. Ωραία. Θα τις πάρουμε λοιπόν επιμέρους. Υπέρ λοιπόν της τροπολογίας 1. Κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 4 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Πάμε τώρα η 76 κατά πίπτη. τροπολογία 7 τώρα. Υπέρ, κατά, υπέρ ξανά, της 7, τροπολογίας 7, υπέρ, Α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 7. Τροπολογία 7. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Με τρεις ψήφους, ε, τέσσερις ψήφους διαφορά. Η Ήτρε 2 καταπίπτει. Τροπολογία 8. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Υπέρ και πάλι παρακαλώ. Κατά Σαφώς εγκρίθηκε. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε η 9. Να ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε την 9 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Καταψηφίστηκε. Είναι σαφές. Συμβαστική τροπολογία 6β. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 78 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Ήτρε 4 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 79 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Οι 12 και οι 5 καταπίπτουν. Τροπολογία 13 τώρα υπέρ. Περ, Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την τροπολογία 13. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Καταψηφίστηκε. Απορρίφθηκε. Ήντα 1 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Είναι σαφές. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Η 14 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η 6 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 15 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 81 υπέρ υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η τροπολογία 82 καταπίπτει η τροπολογία 83 τώρα υπέρ κατά απορρίφθηκε. Γιούρι νομικών υποθέσεων 1 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 85. Απορρίφθηκε η Γιούρι 1, εντάξει. Λοιπόν, η 85 τώρα, υπέρ. 85 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε η 85. Ωραία. Πάμε στην ίντα 2. Σωστό. Ίντα 2 τώρα. Ίντα τροπολογία 2. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές θέλω να πω. Ναι. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 86 καταπίπτει. Ήτρε 8 τώρα. Υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 84 καταπίπτει. Η 87 της κυρίας Ρούλε υπέρ της 87 κατά. Νομίζω ήταν πολύ μικρή η διαφορά. 87 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. επιβραδύνεται ο ρυθμός ψηφοφορίας, πλησιάζει η ώρα του γεύματος, εν πάση περιπτώσει πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε η 87. Τροπολογία 89 τώρα υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε, είναι σαφές. Συμβαστική τροπολογία 5β υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Γιούρι 2 καταπίπτει. Η τροπολογία 20 τώρα υπέρ. Κατά. Συμβαστική Συμβιβαστική τροπολογία 2β υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 91 και ήτρε 10 υπέρ αυτών. Κατά απορρίφθηκαν. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Ήντα 3 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Ήτρε 11 υπέρ υπέρ παρακαλώ, κατά, εγκρίθηκε. Η τροπολογία 23 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. τα 4 υπέρ, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε αυτή. Συμβαστική τροπολογία 8α. Να ψηφιστεί ή είναι ξεχωριστός ο Α, 8α μπεις, υπέρ κατά εγκρίθηκε. Σαφές το αποτέλεσμα. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες 92 και 93. Υπέρ αυτών. Κατά εγκρίθηκαν. Στην τροπολογία 95 και 96 καταπίπτουν. Τροπολογία 24 και 94 καταπίπτουν. Πάμε στην τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. τα Υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. Γιούρι 3 υπέρ κατά και αυτή απορρίφθηκε. Βιομηχανίας 12 υπέρ, ήτρε 12 υπέρ, κατά απορρίφθηκε. Η 98 και η 13 υπέρ αυτών, κατά απορρίφθηκαν. Η 25 υπέρ, κατά εγκρίθηκε. Ήτρε βιομηχανίας 14 υπέρ, κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 25 υπέρ. 26 διορθώνεται. Τροπολογία 26 διορθώνει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Εγκρίθηκε η ΙΤΡΕ 14, γι' αυτό αυτή καταπίπτει, περνάμε στην 27, λέγεται στον πρόεδρο. 27 λοιπόν τώρα, εντάξει, ζητώ συγγνώμη, ε, προχώρησα υπερβολικά γρήγορα και δεν το είδα. 27 υπέρ, εγκρίθηκε 28 υπέρ κατά απορρίφθηκε 29 υπέρ κατά εγκρίθηκε η 99 και μέχρι την 102 υπέρ αυτών κατά απορρίφθηκαν αυτές η 103 υπέρ κατά απορρίφθηκε η 104 υπέρ κατά απορρίφθηκε η 30 υπέρ κατά, εγκρίθηκε. τα 6 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Η 31 τροπολογία υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Η 32 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Η 105 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. τα 7 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Ίντα 8 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Ίντα 9 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Ήτρε 15 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην Ήτρε 16. Ήτρε 16 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 108 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 110 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Είναι τα 10 υπέρ κατά εγκρίθηκε αυτή. Τροπολογία 33 και 34 καταπίπτουν αυτές. Τώρα η τελική ψήφιση του σχεδίου γνωμοδότησης. Άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης της κυρίας Σάντε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και το αποτέλεσμα είναι εγκρίθηκε. 27 ψήφοι υπέρ, 7 εναντίον και 5 αποχές. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Σάντε Μόζε και τους σκιώδους, σκιώδης εισηγητές επίσης για τη συμμετοχή τους. Θέλετε να πείτε κάτι, παρακαλώ. Να πω ευχαριστώ σε όλους για την καλή δουλειά που έγινε. Έχουμε την μεγάλη πλειοψηφία πίσω από την έκθεση, πράγμα σημαντικό για μας για να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Βεβαίως χρειάζεται και το τυπικό βήμα της εντολής. Ελπίζω με βάση το αποτέλεσμα ότι θα έχουμε και εντολή, αλλά θα αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και ευχαριστώ πάλι τους συναδέλφους για αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος αυτού του φακέλου, εποπτεία της αγοράς προϊόντων. Η Αντιπρόεδρος, η κυρία Πιετικάινεν είναι, είναι η συγγήτρια. Θέλετε να πείτε αρχικά δύο λόγια. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και σκιώδεις συγγητές για την καλή και επικοδομητική δουλειά που κάναμε πάνω σε αυτό το θέμα και βεβαίως ε, όλη την υποστήριξη και από τις πολιτικές ομάδες που βοήθησε πάρα πολύ γιατί εν μέρει ήταν πολύ τεχνικής φύσης ο φάκελος αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Είσαστε έτοιμοι για πιο, πολύ, πιο πολλές ψηφοφορίες. Άρθρο 1, παράγραφος 1, ε, ίντα 24. Υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 94 υπέρ κατά απορρίπτεται 95 υπέρ κατά απορρίπτεται 96 υπέρ κατά απορρίπτεται σαφώς 97 υπέρ το 97 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίφθηκε. 98 υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. Όλες απορρίφθηκαν μέχρι τώρα. Είναι 25 υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. 15 του, της εισηγήτριας με προφορική τροπολογία υπέρ κατά δεκτή, 99 κατά πίπτη, είναι 26 υπέρ κατά απορρίπτεται, 100 υπέρ κατά απορρίπτεται. Είναι τα 27 υπέρ κατά απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά απορρίπτεται. 16 της εισηγήτριας υπέρ κατά δεκτή. 102-103 συνδέονται με τη συμβαστική αργότερα. Είναι τα 28 υπέρ κατά απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά δεκτή. Είναι τα 29 πίπτη, 105 πίπτη, συμβαστική 3 υπέρ κατά δεκτή. Πάμε τώρα στην 116 προφορική υπέρ κατά δεκτή. 18 πίπτη, 117 και 118 υπέρ. 117-118 υπέρ κατά απορρίπτονται. 119 και 120 υπέρ κατά απορρίπτονται. 121 υπέρ κατά απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά δεκτή 123 υπέρ κατά απορρίπτεται είναι τα 32 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά δεκτή 5 υπέρ συμβαστική δεκτή και αυτή Πάμε τώρα στην 139 της κυρίας Σαλντεμόζε υπέρ κατά δεκτή, η 123 του εισηγητή είναι τα 35 συμβατή υπέρ κατά απορρίπτεται η 140 υπέρ κατά απορρίπτεται 24 εισηγήτρια υπέρ υπέρ κατά για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό την 24 της εισηγητρίας υπέρ κατά σαφώς δεκτή 141 καταπίπτει είναι τα 36 που είναι συμβατή υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την ίντα 36. Ε, επιταχύνεται λίγο παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. 25 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά δεκτή. 142 υπέρ. Κατά δεκτή. Είναι τα 37 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά δεκτεί. 145 υπέρ κατά απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά απορρίπτεται. 151 και 152 καταπίπτουν. Πάμε στη συμβιβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά δεκτή. Πάμε τώρα στην 158 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 158. Γρήγορα παρακαλώ. Πέρας απορρίπτεται σαφέστατα. Συγγνώμη, δεν είχα δει τα χέρια. 157 υπέρ κατά δεκτή. Είναι τα 39 καταπίπτει, συμβαστική 8 υπέρ κατά δεκτή. Η 9 συμβιβαστική Ίντα 39 λέει είναι συμβατή αν θέλουμε να προσθέσουμε και τα συνδικάτα στην Ίντα 39. Θέλετε να το προσθέσουμε και αυτό ή όχι. Μιλάω για την Ίντα 39 και την προσθήκη End Trade Unions. Πάω πίσω τώρα. Όχι. Όχι λέτε. Ίντα 39. Κατέπεσε το μεγάλο κομμάτι αλλά υπάρχουν και ορισμένες λέξεις που ήταν συμβατές με την 157, ε, που μπαίνουν χωριστά και τα συνδικάτα. Αυτό μπορείτε να το ψηφίσετε. Εγώ σας το επισημαίνω αυτό. Ίσως πρέπει να ψηφίσουμε για να βεβαιωθούμε. Ποιοι είναι υπέρ της προσθήκης αυτών των λέξεων στην 30, από την Ίντα 39. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ωραία. Οπότε είχαμε, είχατε την ευκαιρία να ψηφιστεί. Ψηφίζουμε τώρα την 8. Συμβαστική 8, την ψηφίσαμε αυτή. Την 9 τώρα, υπέρ, κατά, δεκτή. Πάμε τώρα στην 30 της εισηγήτριας, υπέρ, κατά, δεκτή. 166 καταπίπτει, είναι τα 40, είναι συμβατή, είναι τα 40 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 31 υπέρ, της εισηγήτριας υπέρ κατά δεκτή 32 υπέρ κατά δεκτή 167 κατά πίπτη 168 υπέρ κατά δεκτή 169 κατά πίπτη 170 υπέρ ε, Α, θα την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα την 170, μου φαίνεται ότι υπερισσεύει μια σοσιαλδημοκρατική ψήφος. Τώρα είναι καλύτερα. Πέρας. Απορρίφθηκε. Με διαφορά δύο ψήφων. 171 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 172 πίπτη. 173 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 174 υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτή 175 έχει αποσυρθεί 176 υπέρ κατά απορρίπτεται 177 υπέρ κατά απορρίπτεται είναι τα 41 υπέρ κατά απορρίπτεται 178-179 υπέρ κατά απορρίπτονται. 180 υπέρ κατά δεκτή αυτή. 181 υπέρ κατά απορρίπτεται. 33 υπέρ υπέρ κατά δεκτή. Είναι τα 42 συμβατή. Ψηφίζουμε υπέρ κατά Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Ας την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 182. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Σαφώς ναι. Ψηφίζουμε την 183 ως προσθήκη τώρα υπέρ. Κατά δεκτή. 34 υπέρ Κατάδεκτη. συμβαστική 10 υπέρ, κατά δεκτή. Πάμε τώρα στην 188 της κυρίας Ρούλε, υπέρ της 188, κατά, απορρίπτεται, συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά δεκτή. Πάμε τώρα στη 210 με προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 212 καταπίπτει, η 213 είναι συμβατή υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Οι 214 και 215 καταπίπτουν. Α, συγγνώμη, την τα 46. Αυτή θα ψηφίσουμε υπέρ κατά απορρίπτεται 2.14-2.15 είναι κομμάτι της συμβαστικής 11 τη 217 θα ναι, τη 217 υπέρ κατά σαφώς δεκτή 216 έχει γίνει δεκτή λόγω της συμβιβαστικής με, τώρα 218 με το προφορική υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 218 της εισηγήτριας με την προφορική τροπολογία. Πέρας. Δεκτή. Οπότε είναι τα 47 καταπίπτει. Και η 219 καταπίπτει. Οπότε ψηφίζουμε τη 220.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 Ψηφίζουμε τη 220, ελέγχαμε τι καταπίπτει και τι δεν καταπίπτει. 220 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 221 υπέρ, υπέρ, όχι, ηλεκτρονικά θα το ψηφίσουμε αυτό, τη 221 ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με διαφορά τεσσάρων ψήφων ή τριών, λέει ο Πρόεδρος. Η 222 είναι συμβατή με την 221. Την ψηφίζουμε υπέρ. Τη 222 κατά. Απορρίπτεται. 223 και 224 συμβατές επίσης υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 227 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 225 υπέρ κατά, απορρίπτεται. 226 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 228-229 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Είναι τα 48 συμβατή υπέρ, κατά, σαφώς απορρίπτεται. 230-231 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 232-233 υπέρ, κατά, απορρίπτονται 234-235 υπέρ, κατά, απορρίπτονται 236 υπέρ, κατά. Δεν είναι σαφές τι κάνει τώρα το ΕΛΚ εδώ, τη 236. Λοιπόν, ψηφίζομαι υπέρ της 236, κατά, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Δεκτή με τρεις ψήφους. Διαφορά. 237 τώρα, υπέρ. Κατά. Δεκτή. 238 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 239 και 240 μαζί υπέρ κατά δεκτές αυτές ...241-242 υπέρ, κατά δεκτές, 243 υπέρ, κατά δεκτή, 244 ως διαγραφή υπέρ. Υπέρ, κατά, δεκτή. 245 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 245, μου φαίνεται όμως ότι απορρίπτεται. Πιο γρήγορα να ψηφίζετε, λείπουν τρεις ψήφοι. Πέρας. Απερίφθη. Είναι τα 49. Υπέρ. Υπέρ. Πάλι θα ψηφίσουμε και εδώ γιατί είναι παρόμοια τα πράγματα. είναι τα 49. Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Λίγο γρήγορα παρακαλώ. Λοιπόν, έλα, ελάτε, ποιος άλλος είναι, πέρασε της ψηφοφορίας, απορρίφθηκε. Ε, συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, σαφώς ναι, 251 του κυρίου Αρίασα υπέρ, κατά, έλεγχος, συγγνώμη, αλλά ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία, 251 ψηφίζουμε. Ελάτε λίγο πιο γρήγορα παρακαλώ. Πρέπει να κλείσουμε την ψηφοφορία. Ωραία, δεκτή. Εντάξει. 252 καταπίπτει, 40 καταπίπτει, 253 υπέρ. Θα ελέγξουμε πάλι. 253 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε με μια ψήφο. Αποσύρθηκε 254-255 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 257 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 256 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 258 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται 259 και 260 υπέρ κατά δεκτές 262 υπέρ κατά απορρίπτεται 41 υπέρ κατά δεκτή 261 κατά πίπτη 263 υπέρ Α, όχι, θα κάνουμε ένα βήμα πίσω. Τη 261 ως προσθήκη, α, συμφωνεί η κυρία Ρούιλε, η 261 ως προσθήκη, ως προσθήκη τώρα θα την ψηφίσουμε. 261 τώρα ως προσθήκη ψηφίζουμε υπέρ κατά δεκτή. 263 υπέρ κατά απορρίπτεται. 264 υπέρ κατά απορρίπτεται. 265 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά δεκτή, 42 κατά πίπτη, 266 υπέρ, κα, ναι, τη 266, άρχεται η ψηφοφορία επί της 266. Δεκτή. Με διαφορά τριών ψήφων 267 υπέρ κατά απορρίπτεται 268 υπέρ κατά δεκτή 269 υπέρ κατά δεκτή 270 κατά πίπτη, 271 υπέρ κατά απορρίπτεται 272 υπέρ κατά απορρίπτεται 273 υπέρ κατά απορρίπτεται 274 υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτή 275 υπέρ κατά δεκτή 276 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 13 υπέρ κατά δεκτή 284 υπέρ κατά κατά απορρίπτεται 286 υπέρ κατά δεκτή 44 ως προσθήκη υπέρ κατά δεκτή 285 ως προσθήκη υπέρ κατά δεκτή τα 51 υπέρ κατά απορρίπτεται 287 υπέρ κατά δεκτή 288 υπέρ κατά Μπορούμε να ελέγξουμε πάλι για να δούμε. Κατά, κατά ήτανε. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται σαφώς. 291, ε, υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. 289-290 μαζί, υπέρ. Κατά, δεκτές. Οι 45 είναι συμβατή υπέρ, κατά δεκτή. Και οι 292 είναι συμβατή υπέρ, κατά δεκτή. 293 υπέρ, κατά δεκτή. 297 υπέρ, κατά δεκτή. 299 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 300 υπέρ, κατά απορρίπτεται επίσης 301 του κυρίου Αρίας υπέρ κατά 301 του κυρίου Αρίας έλεγχος. Πέρασε. Απορρίφθηκε με διαφορά μιας ψήφου, το ήλεγξα. Ε? Ναι, πρέπει να είστε στην ώρα σας για να ψηφίζετε. Λοιπόν, 303 με προφορική τροπολογία υπέρ. Υπέρ, παρακαλώ. Α, και εδώ πρέπει να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε 303 με προφορική τροπολογία άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Είναι τα 53 υπέρ κατά δεκτή. 302 υπέρ. Καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει. Αφού εγκρίθηκε 53, μάλιστα. Ωραία, ωραία. 302 καταπίπτει. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, πέρασε η ώρα, του βαρυνθήκαμε λίγο. Είναι τα 52 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 304 υπέρ. Κατά. Ε, δεκτή. 305 υπέρ κατά δεκτή, 306 υπέρ, κατά σαφώς ναι. Είναι τα 54 υπέρ, κατά απορρίπτεται. Είναι τα 55 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά δεκτή. 307 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 308 υπέρ κατά απορρίπτεται 47 υπέρ κατά δεκτή 309 υπέρ κατά δεκτή 48 υπέρ κατά δεκτή 310-311 καταπίπτουν 304 του κύριου Φόξ 414 απορρίπτεται, 49 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά δεκτή, 315 υπέρ, κα... α όχι αυτή καταπίπτει, 316 με προφορική υπέρ, κατά δεκτή, 317 υπέρ, κατά δεκτή, 318 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 319 και 320 υπέρ, κατά απορρίπτονται, 321 υπέρ, κατά απορρίπτεται, είναι τα 56 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 323 υπέρ, κατά δεκτή, 322 καταπίτη, 324 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 3.25 και λοιπά υπέρ, κατά απορρίπτονται, 3.28 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 329 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 330 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 331 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 332 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 50 και 3.33 υπέρ κατά δεκτές. 3.34 κατά πίπτη, λοιπόν, 3.35 υπέρ κατά δεκτή. 3.36 υπέρ κατά δεκτή. 338 υπέρ κατά δεκτή. 337 υπέρ κατά δεκτή 339 υπέρ, κατά απορρίπτεται 340 υπέρ, υπέρ παρακαλώ κατά δεκτή 341 την 340 έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 340. Άλλαξε γνώμη το ΕΛΚ. Απορρίφθηκε. 341 υπέρ κατά απορρίπτεται 342 343 υπέρ κατά δεκτές 344 υπέρ κατά απορρίπτεται 345 υπέρ κατά δεκτή και συμβατή 347 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, δεκτή. 346 συμβατή, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 348 ήρθε, 350 υπέρ, κατά, δεκτή και 349 κατά πίπτη. Τώρα είμαστε στο άρθρο 21, 351 υπέρ, κατά, δεκτή. 51 υπέρ, κατά, δεκτή. 353 υπέρ, κατά, δεκτή, 354 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 352 υπέρ, κατά, δεκτή, 355 καταπίπτει, 52 υπέρ, κατά, δεκτή, 356 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 53 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά δεκτή. 360 υπέρ κατά δεκτή. 359 υπέρ κατά δεκτή. 358 υπέρ κατά δεκτή. Συμβατή 54 υπέρ κατά δεκτή. 55 υπέρ κατά δεκτή. Είναι τα 59 συμβατή υπέρ κατά απορρίπτεται. 361 υπέρ κατά απορρίπτεται. 362 υπέρ κατά απορρίπτεται, είναι τα 60 υπέρ, κατά απορρίπτεται, είναι τα 61 υπέρ, υπέρ, κατά απορρίπτεται, 363 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 364 υπέρ, κατά δεκτή, 56 υπέρ, κατά δεκτή, 365 συμβατή υπέρ, κατά δεκτή 57 υπέρ κατά δεκτή είναι τα 62 καταπίπτει 366 υπέρ κατά δεκτή 367 υπέρ κατά δεκτή 369 υπέρ κατά δεκτή 368 συμβατή υπέρ κατά δεκτή 370 υπέρ υπέρ παρακαλώ, της 370 ε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 371 υπέρ, κατά, δεκτή, 372 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 58 υπέρ κατά δεκτή, 374 κατά πίπτη, 375 υπέρ κατά δεκτή, 376 υπέρ, κατά, δεκτή. 377-378 υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τώρα έχουμε την 379 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 380 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 59 της εισηγήτριας υπέρ, κατά δεκτή, 60 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, δεκτή, 381 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 373 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 294 υπέρ, κατά, δεκτή, 295, 296 και 2,98 καταπίπτουν και 3. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά δεξτή. Και πάμε τώρα... Στην 391 άρθρο 33 υπέρ κατά απορρίπτεται. 65 της εισηγήστριας υπέρ κατά δεκτή, 390 υπέρ κατά απορρίπτεται, 389 υπέρ κατά απορρίπτεται, είναι 66 υπέρ κατά απορρίπτεται, 392 υπέρ κατά απορρίπτεται, είναι τα 3 Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι τα 4 υπέρ κατά αποχές δε, απορρίπτεται η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά δεκτή. 12 ε, τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71-73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ευ, απορρίπτονται 72 συμβατή ψηφίζουμε υπέρ της 72 κατά αποχές απορρίφθηκε 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 όχι την είναι τα 9 πρώτα την είναι τα 9 να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, είναι τα 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, είναι τα 11 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται, τροπολογία 2 της εισηγήτριας υπέρ, κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 81 καταπίπτει. Είναι τα 12 συμβατή υπέρ, κατά απορρίπτεται σαφώς, 80 είναι συμβατή, υπέρ, όχι, υπέρ, υπέρ της 80 κατά απορρίπτεται σαφώς 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 14 συμβατή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Είναι τα 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή, 84 συμβατή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 85 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή, είναι τα 17 υπέρ κατά Έλεγχος. Υπέρ της ΣΥΝΤΑ 17. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ώρα είναι να κάνουμε και μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά. Δεκτή. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 20 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε τώρα στη 13 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή 89 και 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, είναι τα 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 91 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, είναι τα 23 υπέρ, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 14, 92, 93 καταπίπτουν και δύο αναφορικέ ε, αναφορικές προτάσεις μαζί να τις πάρουμε. Ε, είναι οι αναφορικές προτάσεις υπέρ και των δύο κατά. Απορρίφθηκαν και οι δύο. Άρχεται η ψηφοφορία η τελική. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε την έκθεση της κυρίας Πιέτη Κάινεν για την εποπτεία της αγοράς. Πέρας. 32 υπέρ 4 κατά, 2 αποχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Φοβούμε ε, ε, πρέπει εδώ ο κύριος Λόκεγκάρντ να μου πει τι πρέπει να κάνουμε. Θέλετε να αναβάλουμε, να το συζητήσουμε το θέμα σας αργότερα. Μπορείτε που θα είναι και περισσότεροι παρόντες. Πότε δηλαδή. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε τώρα. So can Πρόεδρος, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν παρακαλώ να αποχωρήσουν ήσυχα γιατί τις διαφάνειες ε, πρέπει γοργά να μπορέσουμε να τις ε, παρακολουθήσουμε. Λυπούμε Γενική Διεύθυνση GD mark, αλλά περάσαμε πολλή ώρα ψηφίζοντας. Ε. Ποιος είναι που θα παρουσιάσει, θα κάνει αυτή την παρουσίαση. Ησυχία παρακαλώ. Εσείς θα παρουσιάσετε, έτσι. Παρακαλώ. Θα μας παρουσιάσετε λοιπόν. Αλλά βέβαια δεν θα έχουμε χρόνο για πολλές ερωτήσεις, φοβάμαι. Οπότε Ο εισηγητής μας θα παρακολουθήσει τι έχετε να μας πείτε. Και ευχαριστώ και τους διερμηνείς για πέντε λεπτά παραπάνω. Συνεπώς, 8 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας για να μας παρουσιάσετε τις διαφάνειές σας. Έτσι καλώς έχουμε και σε χαρτί τα, τις διαφάνειες αυτές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. 5 λεπτά για το Solvit και το Your Europe. 17 Σεπτεμβρίου εγκρίναμε μία σύσταση και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης. Ο λόγος για τον οποίο θα παρουσιάσουμε μαζί είναι οι επαφές που κάνουμε όσον αφορά τον κύκλο διακυβέρνησης του Solvit που προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα διαφορετικά επίπεδα προκειμένου να λειτουργήσει πραγματικά νομοθεσία για την εσωτερική αγορά. Τι έχουμε κάνει λοιπόν για το Solvit μέχρι τώρα. Στη νέα σύσταση, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη, η οποία ίσχυε από το 2002, έχουμε συμπεριλάβει όλη την πρόοδο που έχει επιταχθεί στο δίκτυο Solvit τα τελευταία 10 χρόνια. Και αν δείτε τον κατάλογο αυτό, εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για μια μικρή εξέλιξη στην δικαιωτική νοοτροπία. Η προηγούμενη σύσταση δεν έλεγε τίποτα για την ποιότητα των υπηρεσιών ή για την πραγματογνωμοσύνη, την νομική ε, το προσωπικό, δεν υπήρχαν αρκετά πράγματα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ποιοτικό έλεγχος ήταν παντελώς απόν και δεν υπήρχε τίποτα για τη συνεργασία με άλλα δίκτυα. Συνεπώς τώρα όλα αυτά καλύπτονται στη σύσταση αυτή, η οποία έχει συζητηθεί με κάθε λεπτομέρεια με τα διάφορα κέντρα Solvit και έχουν εγκριθεί όλα όσα αναφέρονται στη σύσταση. Οπότε αυτό ε, επετέφθη χάρη στο καλό έργο το κέντρο Solvit τα τελευταία 10 χρόνια. Επίσης και χάρη στην συνεχή στήριξη τη δικιά σας, ιδιαίτερα της Επιτροπής ΙΜΚΟ, για την προώθηση του Σόλβιτ και επειδή μας ενθαρρύνατε να πάμε όσο γίνεται πιο μακριά, να προχωρήσουμε πολύ. Τώρα παραμένουν κάποιες προκλήσεις, κάποιες παλιές που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι δεν έχουμε αρκετό ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τον ε, προπολογισμό. Είναι δύσκολο λοιπόν με ταχύτητα να προσφέρουμε υπηρεσίε ποιότητα. Επίση το θέμα του streamlining και εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο ο εξωθρολογισμό δηλαδή των διαδικασιών και επίση, Κάτι άλλο που συνεχίζει να μα απασχολεί είναι ότι πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα προβλήματα τα οποία δεν φτάνουν στο Solvit ποτέ, ιδιαίτερα από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Γιατί αν δείτε αυτό το διάγραμμα που δείχνει τα τελευταία χρόνια τις διάφορες υποθέσεις που έχει επεξεργαστεί το Solvit, θα δείτε ότι το κάτω κομμάτι το μπλε είναι υποθέσεις που έχουν υποβληθεί από τις επιχειρήσεις που παραμένει σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, γιατί οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν το δρόμο για να φτάσουν στο Solvit. Εμεί πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί πολλέ επιχειρήσει δεν είναι ενήμερε για τα δικαιώματά του στα πλαίσια τη εσωτερική αγορά. Εμεί, βέβαια ξέρουμε πολύ καλά τι λέει η νομοθεσία, τα δικαιώματα ε, των ε, καταναλωτών κλπ. Οι επιχειρήσεις όμως δεν τα γνωρίζουν. Και εδώ είναι που έρχεται το Your Europe. Είναι για τους πολίτες, όπως ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχει το κομμάτι δηλαδή Your Europe για τους πολίτες που έχει ε, εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και προσπαθούμε όμως να κάνουμε το ίδιο και για τις επιχειρήσεις. Πριν από λίγες εβδομάδες λοιπόν ξεκίνησε το Your Europe για τις επιχειρήσεις και όπως βλέπετε τώρα παρουσιάζεται με την ίδια μορφή εξίσου φιλικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας συστήνω λοιπόν να πάτε να το κοιτάξετε, να κοιτάξετε αυτή την ιστοσελίδα γιατί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και εδώ είναι που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τα δικαιώματά τους και βάσει αυτού να υποβάλουν τις προσφυγές τους στο Solvit. Θέλω επίσης να τονίσω ότι στις σελίδες Your Europe και στο κομμάτι για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις, σίγουρα χρειάζεται περισσότερη βοήθεια. Κάπου υπάρχει και λέει περισσότερη βοήθεια. Και αν πατήσετε εκεί, τότε βρίσκεται περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη βοήθεια. Αν δηλαδή κάποιο θεωρεί ότι δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του, τότε μπορεί μέσω του Solvit να βρει τη διέξοδο. Στο Your Europe τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι από τότε που ξεκίνησε, το 2010 δηλαδή, έχουμε όλο και περισσότερες επισκέψεις. Φέτος μάλιστα περιμένουμε πάνω από 6 εκατομμύρια επισκέπτες. Είναι πάρα πολύ. Βέβαια δεν μας φτάνει, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά για να είναι ακόμα περισσότερες επισκέψεις αυτές. Γι' αυτό και έχουμε ετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης. Θέλουμε να συμπληρώσουμε το συνολικό πακέτο ενημέρωσης όσον αφορά τις σελίδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καλύψει ένα τμήμα, αλλά περιμένουμε και τα κράτη-μέλη να συμπληρώσουν το δικό τους κομμάτι. Γιατί μπορεί να ξέρει κανείς ποια είναι τα δικαιώματά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν γνωρίζει τι διαδικασίε πρέπει να ακολουθήσει σε εθνικό επίπεδο, τότε θα κολλήσει. Συνεπώ, το πρόγραμμα δράσης εξηγεί τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μπορεί πιο εύκολα να βρει κανείς το Your Europe, να του δώσει μεγαλύτερη προβολή, να το χρησιμοποιεί μέσα από το iPhone ή την ταμπλέτα του ο καθένας και εύκολα να μπορεί να βρει εκεί τις πληροφορίες που ψάχνει. Τα κράτη-μέλη τώρα από τη δικιά τους την πλευρά σε εθνικό επίπεδο πρέπει να δώσουν περισσότερες πληροφορίες, να φροντίσουν για links με εθνικές πύλες, μέσω δηλαδή εθνικών πυλών προς το Your Europe να υπάρχει επίσης και μεγαλύτερη διαφήμιση. Υπάρχει μια ε, σελίδα Facebook που έχει αναλάβει ένας από τους συναδέλφους μας. Εμείς διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στο Twitter αναφέρουν πράγματα για το Your Europe και συστήνουν ο ένας τον άλλον να επισκεφθούν το Your Europe. Οπότε γι' αυτό θα ήθελα και εσείς αν έχετε λογαριασμό Twitter αναφέρεται το Your Europe σαν ένα, ένα σημείο στο οποίο μπορεί να πάει κάποιος για να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του. Τέλος, αν θέλετε συνολικά να ξέρετε τι γίνεται όσον αφορά την διακυβέρνηση, πηγαίνετε στο online βαθμολόγιο για την εσωτερική αγορά και θα βρείτε πολύ περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση όσον αφορά την Ευρώπη, το Solvit, αλλά και ως σημείο ενιαίας επαφής. Τέλος, ένας κατάλογος με links όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα όσα σας ανέφερα μέχρι τώρα. Και για να τελειώσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην Επιτροπή ΙΜΚΟ για την συνεχή σας στήριξη προς το Solvit και το Your Europe. Νομίζω ότι η στήριξη αυτή έκανε τη διαφορά. Έχουμε προχωρήσει πολύ. Εννοείται ότι μένει ακόμα αρκετής δρόμος. Γι' αυτό θέλω να σας ζητήσω να συνεχίσετε στον ίδιο ρυθμό και να φροντίζετε, με ένα πάσα στιγμή, κάθε φορά που σας δίνεται η ευκαιρία, να αναφέρετε το τους στους πολίτες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη σαφή και πλήρη ενημέρωση που μας δώσατε. Ναι, τις διαφάνειες οδός θα τις δώσουμε σε όλους τους ευρωβουλευτές και όλα αυτά που είπατε για το Twitter κλπ. Ένα λεπτό εισηγητής, παρακαλώ. Σε ένα λεπτό, ναι. Συστήνω Όντω να δίνουμε στον κόσμο πέντε λεφτά και τότε θα μπορούμε να έχουμε πάντα τόσο εξαίρετε παρουσιάσεις όπως και αυτή που μόλις ακούσαμε. Υπογραμμίζεται λοιπόν εδώ η κατάσταση πραγμάτων και αναφέρονται οι συστάσεις για το πώς θα φέρουμε το Solvit στο επόμενο επίπεδο. Όπως μόλις ακούσαμε, έχουμε δύο εκθέσεις. Έχουμε τις συστάσεις των αρχών όσον αφορά τις χώρες μέλη και μετά έχουμε το Your Europe για τους πολίτες και ε, τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι και οι δύο αυτές εκθέσεις παρουσιάζουν πολύ καλά τη σημερινή κατάσταση. Βέβαια, τίθεται και διάφορα που αναφέρει η έκθεσή μου και θα ήθελα να τα κοιτάξετε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε γενικά το σύστημα. Λειτουργεί όπως θα θέλαμε να λειτουργεί. Δεύτερον, ποιος χρησιμοποιεί τελικά το δίκτυο Solvit. Όπως είδαμε, αρχικά πρόθεση ήταν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις να το χρησιμοποιούν. Όμως, διαπιστώνουμε, το είδαμε μόλις, ότι κυρίως οι πολίτες χρησιμοποιούν το Solvit. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ώστε να έχουν περισσότερες επιχειρήσεις πρόσβαση στο Solvit, να απευθύνονται σε αυτό πιο πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχουν εμπόδια και μου το έχουν πει και από το Solvit και οι επιχειρήσεις. Χωρίς όμως να ξέρουμε τελικά αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή, πού οφείλεται αυτό τελικά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε περισσότερο στην έκθεση. Αναφέρθηκε το θέμα της προβολής του Solvit, της ενημέρωσης του κόσμου γι' αυτό. Είναι περιορισμένα. Γιατί εσείς λέτε ότι είναι ένα πρόβλημα, αλλά και πριν από τέσσερα χρόνια ήταν. Και βέβαια να δούμε και το νομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να ετοιμάσει το νομικό πλαίσιο της διακυβέρνησης του Solvit και εκφράζω την ικανοποίησή μου γι' αυτό στην εκθεσή μου. Τέλος, τα κράτη-μέλη. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Το αναφέρετε και εσείς αυτό. Συνεπώς, πρέπει να φέρουμε το Solvit στο επόμενο επίπεδο πρέπει να έχουμε την επόμενη εκδοχή. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Πρόεδρος, πρέπει να ολοκληρώσουμε, οπότε φοβάμαι πως οι σκιώδεις δεν θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουν. 8 Νοεμβρίου περιμένουμε την έκθεσή σας. Επίσης υπάρχει δικιά μας η έκθεση, έτσι, για το ενιαίο Ευρωπαϊκό Σημείο Επαφής. Υπάρχει στην ιστοσελίδα. Ο εισηγητής θα το αναφέρει δίχως άλλο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα τους εισηγητές που καταφέραμε σε τόσο λίγο χρόνο να το συζητήσουμε. Προσβλέπω σε επόμενες συζητήσεις μας για αυτό το θέμα. Τρεις η ώρα θα συνεχίσουμε εδώ. Ευχαριστώ.